Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Έχουμε λίγο λιγότερο από 45 λεπτά, 40 λεπτά για την συνεδρίασή μας. Για να εκμεταλλευτούμε και την παρουσία των διερμηνέων που τους ευχαριστώ και για την τεχνική συζήτηση που είχαμε πριν. Έχουμε το πρόγραμμα Δικαιοσύνης. Θα ήθελα να χαιρετήσω την παρουσία του κυρίου Βάιντεν Χόλτσερ που εκπροσωπεί την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και είναι και συνεισηγητής του θέματος αυτού. Θα σας πρότεινα ο καθένας να πάρει το λόγο για 15 λεπτά και κατόπιν θα εξαντλήσουμε τον υπόλοιπο χρόνο. Καταρχήν η κυρία Χαουτάλα όμως έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η συνεργασία με τον συνσηγητή, τον κύριο Βάιντεν Χόλτσερ, ήταν εξαιρετική και πρόσκοπτη. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το σχέδιο της έκθεσης. Θα πρέπει να ξέρετε, αυτό το πρόγραμμα είναι παράλληλο με το πρόγραμμα των δικαιωμάτων και των αξιών, το οποίο παρακολουθούμε επίσης για να διασφαλίσουμε ότι συμπληρώνει το ένα το άλλο και ότι και τα δύο αποτελούν το Ταμείο για τα Δικαιώματα και τις Εξίες στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων επίσης γνωμοδοτεί για ε, τη ΛΥΜΠΕ για το πρόγραμμα για τις αξίες και τα δικαιώματα για το οποίο αρμόδια είναι η ΛΥΜΠΕ. Το πρόγραμμα δικαιοσύνης μας δίνει εξαιρετικές ευκαιρίες ε, να δούμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε την κατάρτιση των επαγγελματιών ε, στο νομικό κλάδο και τα δίκτυα και πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τα δίκτυα ε, των διάφορων οργανισμών υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των Ombudsman, των ιδρυμάτων κατά της εισαγωγής διακρίσεων κτλ. Το σημαντικό είναι πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την πρόσβαση, να διευκολύνουμε την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τα θύματα, ένα ιδιαίτερα επώδυνο ζήτημα, το οποίο δεν το αντιμετωπίζουμε όπως πρέπει. Ε, γι' αυτό τέτοια δεσυνοριακά εγκλήματα όπως η εμπορία ανθρώπων ε, αναφέρονται στις τροπολογίες μας. Γιατί αν δείτε την εμπορία ανθρώπων είναι ε, ουσιαστικά με από τις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις σήμερα παγκοσμίω και τα θύματα λόγω της δεσυνοριακής φύσης των εγκλήματων αυτό είναι πολύ σημαντικό να αναπτύξουμε μέσα για να βοηθήσουμε τα θύματα και να αντιμετωπίσουμε αυτά τα εγκλήματα. Νομίζω αυτά χρειάζεται να πω. Να προσθέσω όμως ότι με τον ε, συνεισηγητή θέλουμε το παράρτημα 1 να εισακθεί στο διατακτικό του νομοθετήματος, γιατί αυτό θα προσέθεται σαφήνεια. Δεν βλέπουμε κανένα λόγο το παράρτημα 1 ε, να μην είναι μέρος του νομοθετήματος. Ενώ το παράρτημα 2 που αφορά τους δείκτες θα μπορούσε να παραμείνει ως παράρτημα. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τη σαφήνεια και τη συντομία. Τώρα ο κύριος Βάιντεν Χόλσερ. Σας ευχαριστώ θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω θερμά τη συνεισηγήτρια για την καλή συνεργασία που είχαμε. Ήδη ανέφερε ότι έχουμε να κάνουμε εδώ μια προγράμματα. Ε, το πρώτο το οποίο είχε συζητηθεί από την Επιτροπή ΛΥΜΕ και το άλλο, το πρόγραμμα δηλαδή δικαιοσύνης. για τα οποία προγράμματα βέβαια έχει προβλεφθεί το ίδιο ποσό των χρηματοδοτικών κοντιλίων όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Και βέβαια η δική μου πρόταση από κοινού με την Χάιντι αλλά είναι ότι θα πρέπει να αυξηθούν τα εν λόγω κονδύλια. Επίσης το ζητούμενο είναι να τονίσουμε, να δώσουμε περισσότερη έμφαση στο ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και έχουν υποβληθεί σχετικέ τροπολογίες από τη μας πλευρά. Προτείνονται τροπολογίες. Επίσης, ο στόχος μας είναι να αναφερθούμε και στον ρόλο του κράτους δικαίου για σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Δηλαδή να γίνει αυτή η προσθήκη του κράτους δικαίου. Επίσης, Επίσης αναφερόμαστε στην ανάγκη της ε, ανταλλαγής απόψεως στην κοινωνία των πολιτών, ενός διαθρωμένου δηλαδή διαλόγου ε, της κοινωνίας των πολιτών, structured civil dialogue. Και επίσης η διάρκεια του προγράμματος δεν θα πρέπει να είναι τέσσερα χρόνια όπως προτείνει η Επιτροπή, αλλά δύο γιατί θεωρούμε πως έχει περισσότερο νόημα να έχει μικρότερο βάθος χρόνο έτσι ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε ενδεχόμενε αλλαγέ τις οποίες ε, μπορούμε να προβούμε. Δηλαδή, μέσα στα δύο πρώτα χρόνια να μπορέσουμε να κάνουμε τις ε, πρώτες τροποποιήσεις αν χρειαστεί στο σύνολο των 7 συνολικών ετών του προγραμματος. Τώρα, σε ό,τι αφορά την προθεσμία για την υποβολή των τριπολογιών είναι 5η Δεκεμβρίου. 5 Δεκάτου. Μετά έχουμε βέβαια το διάλειμμα αυτό των Χριστουγέννων και μετά η δεκεμβριου 5 Δεκεμβρίου. μετα εχουμε βεβαια το διαλειμμα τροπολογιών θα γίνει 23 και 24 Ιανουαρίου. Η ψηφοφορία τώρα στις αρμόδες επιτροπές θα λάβει χώρα αρχές Φεβρουαρίου έτσι ώστε να ψηφιστεί ε, πρόταση το Μάρτιο στην Ολομέλεια, δηλαδή πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του τρεχόντου Συνοβουλίου. Αυτά λοιπόν είναι πρόσθετων σχολείων στα όσα είπε η συνάδελφος Να Ευχαριστώ πολύ. Ποιος θέλει το λόγο. πιστεύω. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Οι ε, δύο ε, δική μας της από το ΕΛΚ δεν ε, κατάφεραν να παρευρεθούν, οπότε ε, θα σας διαβάσω κάτι τη πλευρά. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, σκιώδεις, οι μας λοιπόν, άδευ και ΔΙΔΙΕ είναι έκπληκτη με το γεγονό ότι κανένα από τα σχόλια που έκαναν κατά την αρχική ανταλλαγή απόψεων ε, ε, με την ΟΠΗ δεν ελήφθησαν υπόψη. Ειδικότερα το σχόλιο που έκαναν σε ό,τι αφορά ε, την ανεξαρτησία των δικαστών. Το σχέδιο της έκθεσης, έτσι όπως παρουσιάζεται, παρεκκλίνει σοβάρα από τον στόχο του προγράμματος δικαιοσύνη, που είναι η ενίσχυση των εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης των κρατών μελών ενώ περιλαμβάνει αυτή η πρόταση έκθεση ε, ε, ε, σε οι οποίες έρχονται σε, αρχές, σε, σε, αντίθεση με τις αρχές σε ό,τι αφορά ειδικότερα το ρόλο τη κοινωνία των πολιτών και επίσης άπτονται της πρότασης που έχει γίνει σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με γενικότερες έλευσεις και το κράτος δικαίου στα κράτη-μέλη. Η, η διεύρυνση του ορισμού ε, του δικαστικού σώματος έτσι ώστε να περιλαμβάνει τους νομικούς εμπειρογνώμονες, της οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, ε, οι συγκεκριτέ μας θεωρούν πως είναι αρκετά προβληματικό. Γι' αυτό αντί να δημιουργήσουμε τελικά ένα συνακτικό νομικό πλαίσιο για την ε, περίοδο 2021 έως 2027, τελικά ενδέχεται να οδηγηθούμε σε μια κατάσταση όπου έχουμε αλληλευκολεπτόμενα προγράμματα και νομοθεσίες, εάν ακολουθήσουμε την προσέγγιση μας προτείνουν οι εισηγητές. Κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο ε, για το έλεγε, γιατί ουσιαστικά θα οδηγήσει σε διασπάθηση ενωσιακών κονδυλίων. Επίσης, η τροπολογία 17 σε ό,τι αφορά την πρόσβαση της δικαιοσύνης, ε, θεωρούμε πως είναι υπερβολικά ευρεία γιατί ένα άρθρο ενός κανονισμού ουσιαστικά μεταβάλλεται σε μια πολιτική δήλωση, πράγμα το οποίο από νομικοτεχνικής άποψης ε, δεν είναι ορθό. Επίσης, η τροπολογία 18 είναι υπερβολική γιατί υπερβαίνει τα όσα ήδη προβλέπονται μέσα στην ενωσιακή νομοθεσία. Εμείς λοιπόν θα υποβάλουμε τροπολογίες οι οποίες πραγματικά μπορούν να βοηθήσουν τα εθνικά συστήματα δικαιοσύνης των κρατών μελών με στόχο την ενίσχυση της ανεξαρτησίας τους και της άμερολεψίας τους ανταποκρινόμενοι στι απαραίτητες προσαρμογές τους στις ε, νέες προκλήσεις και στις αλλαγές που υπέρχονται και με την ε, νέα ενωσιακή νομοθεσία. Κάφμαν. Κύριε Κάφμαν. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Πρόεδρε. Ίσως ε, βέβαια να μην εκπλαγεί ο κύριος Φως αλλά μετά από την δρυμία κριτική που άσκησε στην πρόταση, εγώ θα ήθελα να πω ακριβώ το αντίθετο. Δηλαδή ότι επιχαίρω αυτή την έκθεση, το σχέδιο έκθεση ε, των συναδέλφων Βέντεν Χόλτσα και Άουταλα, γιατί πραγματικά θεωρώ πω ε, ε, σε αυτή την έκθεση θίγουν πολύ σημαντικά ζητήματα, όπω για παράδειγμα η διατήρηση του κράτου δικαίου, γενικά η τήρηση των νόμων στα κράτη-μέλη πράγμα το οποίο νομίζω πως θεωρούμε όλοι μας πως αποτελεί βάση για την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών και την εμπιστοσύνη στα νομικά συστήματα των άλλων κρατών μελών καθώς βέβαια ε, απαραίτητη προϋπόθεση για αυτή την εμπιστοσύνη είναι η αμεροληψία των ε, δικαστών. Και φυσικά, εάν μια τέτοια τροπολογία από την πλευρά του ΕΛ και θέλει να δώσει περισσότερη έμφαση σε αυτή την αμεροληψία, το ορίζουμε. Ένα δεύτερο στοιχείο που ε, αναφέρουν σωστά οι συζητές είναι περαιτέρω ε, μέτρα για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη ε, προ όφελο των θυμάτων παρανόμων πράξεων. Δηλαδή συχνά κάνουμε λόγο εδώ για αδικήματα, για το τι θα πρέπει να γίνει προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών, αλλά συχνά δεν λαμβάνουμε υπόψη μας τη διάσταση του θύματος, την οπτική αγωνία του θύματος. Και γι' αυτό θεωρώ πως ε, πραγματικά αυτό το σημείο που θίγουν οι συγκητές είναι πολύ χρήσιμο. Επίσης η πρόταση οι οργανώσεις εκείνες της ε, κοινωνίας των πολιτών που ενδιαφέρονται ακριβώς και υπερασπίζονται τα δικαιώματα των θυμάτων ε, να λαμβάνουν κάποια κονδύλια στο μέλλον είναι κάτι το οποίο υποστηρίζουμε. Ένα τρίτο στοιχείο που μας αρέσει και που εκφράζεται στο, στην έκθεση Ε, είναι ότι θα πρέπει όσοι κάνουν τις σχετικές αιτήσει και οι συμμετέχοντες ε, να εστιάζουν ακριβώς στο έργο που επιτελούν στο πλαίσιο του προγράμματος. Δηλαδή θα πρέπει να ε, είναι ελάχιστη η διοικητική τους επιβάρυνση καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, δηλαδή από την υποβολή της αίτησης μέχρι την εκταμίευση. Και τέλος, να κάνω και ένα τελευταίο σχόλιο για να γνωρίζει ο κύριο Φώσο ότι τον άκουσα προσεκτικά. Και αυτό είναι το εξή. Έχουμε δύο προγράμματα, το πρόγραμμα για τη δικαιοσύνη και το πρόγραμμα για τα δικαιώματα και τις αξίες και πράγματι ναι θα πρέπει να προσέξουμε να μην υπάρξει άλλη λεπικάλυψη μεταξύ των δύο προγραμμάτων δηλαδή να προσέξουμε να τα οριοθετήσουμε και να ξέρουμε γιατί προβλέπεται το ένα και γιατί το άλλο είμαι σίγουρος ότι οι συγκητές θα το λάβουν αυτό υπόψη τους. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστώ. κυρία Κινίτση έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως και η συνάδελφος Κάφμαν θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Χάουταλα και τον συνεισηγητή της για μια εξαιρετική προσπάθεια γύρω από τα θέματα της δικαιοσύνης. Ε, ήμουν σκιώδης εισηγήτρια στα θέματα αυτά και γι' αυτό θα ήθελα να ε, αναφερθώ εκ νέου σε αυτά τα οποία τέθηκε ε, στα προβλήματα τα οποία τέθηκαν. Ήμουνα και δικαστής πριν έρθω εδώ και γνωρίζω αρκετά για την ανεξαρτησία, τη σημασία της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και τη σωστή συνεργασία ανάμεσα στα διάφορα επαγγέλματα στον τομέα της δικαιοσύνης. Κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για τη σωστή διαχείριση της δικαιοσύνης. Και γι' αυτό ακριβώς το πρόγραμμα αυτό για τη δικαιοσύνη έχει προσφέρει ιδιαίτερα δημιουργώντας τα λεγόμενα διεθνικά δίκτυα, τα οποία έχουν σαν στόχο την κατάργηση, την κατάρτιση συγγνώμη, των δικαστών και στον αστικό τομέα και στον ποινικό, όπως επίσης και στην αναγνώριση των δικαιωμάτων των θυμάτων. Νομίζω ότι πρέπει το θέμα αυτό να αποτελέσει μια προτεραιότητα για το επόμενο πρόγραμμα 21-27 και αναφέρθηκε σε αυτό η κυρία Κάουφμαν ε, στην περίπτωση των θυμάτων σε περιπτώσεις διασυνοριακές και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί και θα εξεταστεί και από την Ειδική Επιτροπή για την Τρομοκρατία της οποίας είμαι μέλος. Ε, σχετικά τώρα με τα δικαιώματα και την προστασία των ανηλίκων. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει έτσι ώστε να εκπαιδεύονται σωστά και οι δικαστές και οι δικηγόροι και όσοι ασχολούνται με θέματα των ανηλίκων γενικότερα. Όπως επίσης και η προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων που εμπλέκονται σε ε, ποινικέ και σε δικαστικές μάλλον ε, διαδικασίες γενικότερα. Και υπάρχει και το θέμα επίσης των ανηλίκων που ζουν ε, κάτω από συνθήκες δύσκολες στην περίπτωση που οι γονείς τους βρίσκονται σε σοφρονιστικά καταστήματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε, είναι θέμα θα έλεγα ανθρωπισμού το να δούμε τις συνθήκες κράτησης είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να μην αντιμετωπίσουμε στο επόμενο πρόγραμμα για τη δικαιοσύνη 21-17. Σας ευχαριστώ όλους για την καλή σας προσπάθεια και θα προσπαθήσω και εγώ να συνεισφέρω στο τελικό κείμενο σε συνεργασία με τους υπόλοιπους σκιώδεις και συντονιστές. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κινίτσι. Γερεκ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την προηγούμενη ομιλήτρια για τα θέματα τα οποία έθεσε, ιδιαίτερα το θέμα της προστασίας των θυμάτων αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να ανήκει, θα έλεγα, σε μια τέτοια έκθεση. Βέβαια υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία μας ανησυχούν εδώ. Αναφέρομαι στα θέματα της δικαιοσύνης, αλλά το να εντάξουμε την ε, σύμβαση της Κωνσταντινούπολης δεν είναι κάτι το οποίο θα έλεγα θα προκαλέσει μια κάποια σύγχυση στις συζητήσεις που γίνονται στα κράτη-μέλη γιατί ξέρετε ότι πολλές χώρες, ιδιαίτερα στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, δεν έχουν επικυρώσει τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και μάλιστα το δικαστήριο στην Βουλγαρία έχει αποκλείσει κάθε μορφή επικύρωση της ε, σύμβασης αυτής. Ε, γιατί υπάρχουν ε, αντιθέσεις με την έννοια ας πούμε ε, οικογένεια στο βουλγαρικό δίκαιο. Συνεπώς λοιπόν δεν θα πρέπει να απευθύνουμε εκκλήσεις για να παραβιάζονται οι αποφάσεις των ανωτάτων δικαστικών αρχών. Έχουμε να κάνουμε με δημοκρατικές χώρες και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιο μόντος βιβέντη έτσι ώστε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μεταξύ μας και να μην προσπαθήσουμε η πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιβάλλει τις θέσεις της στην μειοψηφία. Επίσης έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του προγράμματος αυτού, οι οποίες δεν έχουν ακόμα αποδώσει. Αν υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία δημιουργούν αμφιβολίες και αντιθέσεις, δεν μπορούμε εμείς να στηρίζουμε τη μία πλευρά εις βάρος της άλλης έτσι εύκολα, γιατί η φιλελεύθερη δημοκρατία μας στην περίπτωση αυτή διατρέχει τον κίνδυνο να καταστεί μη φιλελεύθερη. Υπάρχουν λοιπόν χώρες οι οποίες ε, όταν υπάρχουν προβλήματα πολιτικά ανάμεσα σε χώρες ε, μπορούν να στηρίξουν τη μία πλευρά εις βάρος της άλλης, αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι υπέρ της δημοκρατίας γενικότερα. Εμείς δεν θέλουμε λοιπόν η έκθεση να ασχολείται με τέτοια διφορούμενα θέματα. Θέλουμε να καταστήσουμε την έκθεση πιο λειτουργική και πιο διαφανή. Και θέλουμε να καταστήσουμε επίσης και πιο α, σαφείς ε, στόχους των δύο προγραμμάτων. Εμείς λοιπόν σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει ε, να υπακούμε στις ευρωπαϊκές συνθήκες πριν από οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν πολλά θέματα, οι προηγούμενοι ομιλητές αναφέρθηκαν στα θέματα αυτά και θα πρέπει πριν από οτιδήποτε άλλο να σεβαστούμε την αρχή της επικουρικότητας και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να παρεμβαίνουμε στις νομικές διαδικασίες κάθε χώρας. Σας ευχαριστώ κύριος Λεμπρετό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το κείμενο το οποίο έχουμε μπροστά μας σήμερα είναι σημαντικό κείμενο το οποίο έχει σχέση με το πρόγραμμα δικαιοσύνη και έχει σαν στόχο να βελτιώσει την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα των κρατών μελών. Στο σχέδιο το οποίο έχουμε μπροστά μας υπάρχουν θα έλεγα αρκετά ενδιαφέρουσες προτάσεις. Οι τροπολογίες 2, 18 σχετικά με την περιβαλλοντική εγκληματικότητα ή σχετικά με τη σώματεμπορία. Είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και η ιδέα η οποία περιλαμβάνεται στην τροπολογία 28 ότι θα πρέπει να υπάρξει ειδική προστασία στα θύματα σε περιπτώσεις διασυνοριακές προφανώς είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό και πρέπει να μας απασχολήσει. Πέραν τούτου όμως, αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση στην έκθεση αυτή είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές τροπολογίες για την υποστήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό με τρομοκρατεί, γιατί οι οργανώσεις αυτές, οι ΜΚΟ, δεν θα πρέπει να φανούμε συναισθηματικοί, δεν είναι οργανισμοί που τείνουν να βελτιώσουν τη δικαιοσύνη, είναι οργανισμοί που τείνουν να αποσταθεροποιήσουν πολιτικά καθεστώτα και να κάνουν επεμβάσεις στις εσωτερικές υποθέσεις χωρών. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες γύρω από αυτήν την υπόθεση αυτή η 19 σαν παράδειγμα η οποία λέει ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις ΜΚΟ όπως επίσης και η 29, 32 και 38. Εγώ διαπιστώνω ότι εδώ υπάρχει μία θα έλεγα αντίληψη αρνητική. Και υπάρχει και κάτι άλλο που με απασχολεί, η αναφορά που γίνεται στα πλαίσια της τροπολογίας 29 στην λεγόμενη καθολική δικαιοδοσία. Ίσως εδώ να υπάρχει θέμα μετάφρασης αλλά αν είναι αναφορά στην λεγόμενη έννοια της παγκόσμιας δικαιοσύνης που επιτρέπει σε οποιαδήποτε χώρα να κρίνει οδήποτε έγκλημα σε μια άλλη χώρα, τότε εγώ φυσικά και είμαι εναντίον. Δεν θέλω την έννοια αυτή της, της δικαιοσύνης γιατί είναι μέσω των ισχυρών χωρών να παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις των ασθενέστερων. Εγώ είμαι υπέρ της χάρτας των Ηνωμένων Εθνών που λέει ότι η δικαιοσύνη είναι ίση σε όλες τις χώρες. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Θα ξαναδώσουμε το λόγο για καταληκτικέ παρατηρήσεις ε, στους ε, συνσηγητές, αλλά να ρωτήσω και την Κομισιόν μήπως ε, θέλει το λόγο. Ναι ή όχι. Πιστεύω πω ναι. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να εκφράσω άποψη, απλώς να ευχαριστήσω τους δύο συγγητές για την έκθεση και να απαντήσω και σε κάποια σχόλια που έγιναν το σημείο δηλαδή το γεγονό ότι έχουμε δύο προγράμματα που χρηματοδοτούνται από ένα ταμείο και είπατε ορθά ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει συμπληρωματικότητα μεταξύ των δύο προγραμμάτων, θα πρέπει να αναπτυχθούν συνέργειες μεταξύ των δύο προγραμμάτων που προκύπτει ότι γεγονό ότι το πρόγραμμα για τη δικαιοσύνη θα διαφέρει από το σημερινό σε κάποιο βαθμό, αλλά ταυτόχρονα ισχύει ότι θα πρέπει να αποφύγουμε και τις επικαλύψεις. Όμως, όπως υπόθηκε στο γεγονό ότι και η Επιτροπή λιμπεργάζεται εργάζεται επί των δύο προγραμμάτων, αποτελεί εγγύηση ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τα δύο προγράμματα λοιπόν θα πρέπει να συμβαδίζουν. Και ένα άλλο σημείο αφορά τις ε, δραστηριότητες που μπορεί να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα αυτό. Μιλάμε για ευρία γκάμα δραστηριοτήτων και επίσης και για μεγάλη γκάμα δικαιούχων. Αν ε, το συγκρίνουμε με το πρόγραμμα για τα δικαιώματα και τις αξίες, η ιδιαιτερότητα του προγράμματος για τη δικαιοσύνη είναι πως αν δείτε τον κατάλογο των δραστηριοτήτων, ε, κάποιες ε, δραστηριότητες ε, ουσιαστικά είναι στα μέτρα κάποιων δικαιούχων. Πρέπει το χάρη η κατάρτιση, η δικαστική απευθύνεται στους δικαστές και στο δικαστικό προσωπικό και άλλες δραστηριότητες που απευθύνονται στις ΜΚΟ. Εδώ έχουμε διαφοροποίηση με το πρόγραμμα δικαιωμάτων και αξιών, γιατί έχουμε πιο εγκάρσια κατανομή των δραστηριοτήτων, αν θέλετε. Επίσης, υπήρξε ένα σχόλιο για τα δύο έτη παρακολούθησης. Θέλω να αποσαφηνίσω ότι δεν μιλάμε για τήσια παρακολούθηση, γιατί θα κάνουμε την παρακολούθηση ένα έτος, αλλά εδώ μιλάμε για την ενδιάμεση αξιολόγηση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα του προγράμματος για να κάνουμε μία πλήρη μελέτη. Και υπάρχει διοργανική συμφωνία της καλύτερης νομοθεσίας που λέει ότι τουλάχιστον θα πρέπει να έχουμε δεδομένα τριών ετών, πλήρη δεδομένα, για να κάνουμε μία σωστή αξιολόγηση. Και όταν ε, τρέχουμε προγράμματα θα πρέπει να παρουσιάσουμε ε, τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, θα πρέπει να λάβουμε τις απαντήσεις. Αυτά λέει η Οργανική Συμφωνία, αλλά εδώ δεν μιλάμε για την παρακολούθηση. Η παρακολούθηση γίνεται ετησίως. Εδώ συμφωνούμε μαζί σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και τις διευκρινήσεις σας. Τώρα να περάσουμε στις τελικές παρατηρήσεις των δύο συγητών. Θα ξεκινήσουμε τον κύριο Φάιντεν Χόλτσερ. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ε, παρατηρήσεις που κάνατε και οι οποίες εν μέρη ήταν θετικές. Αλλά θα ήθελα να ε, πω ότι θα επανεξετάσω και τα επικριτικά σχόλια που ακούστηκαν. Γιατί σίγουρα μπορούμε ε, να μάθουμε περισσότερα από την κριτική από, τη, από τους επένους. Οπότε με βάση αυτή την κριτική θα προσπαθήσουμε να ε, επανεξετάσουμε την έκθεση έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη μας αυτά τα σημεία. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά δηλαδή τις τροπολογίες εκείνες για τις οποίες θα ασκηθεί γενικότερα κριτική. Καθώς ε, λέτε κύριε Βεντενχόλσερ ότι οι κριτικές είναι πιο χρήσιμες από τους επένους, ε, εδώ ξέρετε ότι είμαστε πολύ ακριβείς στην κριτική και ε, πολύ φιδωλοί σε επένους. Η κυρία Χαρτάλα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ενδιαφέρον να, να ακούμε ότι εμείς οι δύο δεν θα πρέπει καθόλου να φύγουμε τέτοια πολύ σημαντικά θέματα που είναι εξαρτησία των δικαστών. Φυσικά και πρέπει να το κάνουμε μέσω της κατάρτισης ε, των επαγγελματιών στον κλάδο της δικαιοσύνης και αναφερόμαστε και στην κατάρτιση των δικαστών και των λοιπών επαγγελματιών. Έτσι λοιπόν, με εκπλήσει το ότι στην πρόταση της Κομισιόν ούτε στις τροπολογίες μας δεν βρίσκουμε αυτή τη βασική προσέγγιση που θα πρέπει να αφορά όλους τους επαγγελματίες του κλάδου, θα πρέπει να σέβονται την ε, όλες τις αρχές του κράτους δικαίου και φυσικά η ανεξαρτησία των δικαστών είναι κλειδί. Επίσης, ε, ακούσαμε μια κριτική από τον κύριο Ντιτιέ για το θέμα της κοινωνίας των πολιτών. Βέβαια, από το στόμα του κύριου Φως. Νομίζω ότι υπάρχει παρεξήγηση. Δεν προσπαθούμε να πούμε ότι η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να παίξει το ρόλο των δικαστών ή των εισαγγελέων ή κάτι τέτοιο. Αλλά ξέρετε ότι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη είναι ένα θέμα κλειδί το να λειτουργεί το δικαστικό σύστημα και το κράτος δικαίου. Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν πρόσ... που θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη δεν είναι πάντοτε σε θέση να φτάσουν στη δικαιοσύνη. Γι' αυτό αποφασίσαμε να δώσουμε έμφαση και στο ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στο πώς θα βοηθήσει για να αναπτυχθούν ε, κάποιες ε, υποθέσεις διαφορών για τα θύματα και για όσους θα πρέπει να γνωρίζουν πώς μπορούν να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Επίσης με εκπλήσει που υπήρξε τόση κριτική ο κ. Λιμπρετών παραδείγματος χάρη μπορεί να κατάλαβα γιατί δεν θέλετε να δούμε τίποτα για την καθολική δικαιοδοσία, για την παγκόσμια δικαιοδοσία. Όμω είναι αλήθεια ότι τα νομικά μα συστήματα αναπτύσσουν και αυτή την αρχή τη παγκόσμια δικαιοδοσία. Θα πρέπει να σκεφτείτε τις γυναίκες γεζίδη που ήταν θύματα του Άισι στο Ιράκ και στη Συρία. Πιθανότατα, ο μόνος ε, τρόπος να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα θύματα αυτά είναι μέσω της παγκόσμιας δικαιοδοσίας. Πολλές χώρες ε, ήδη προβαίνουν στην άσκηση τέτοιας δικαιοδοσίας. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό, όπως προσπαθήσαμε να κάνουμε, να τονίσουμε τη δυσκολία του διασυνοριακού στοιχείου των αξιόπινων πράξεων που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Και αυτό σημαίνει και πάλι κατάρτιση για τους επαγγελματίες του κλάδου. Μια άλλη δυσκολία για την άσκηση της δικαιοσύνης σήμερα είναι διάφορες ε, πολυπλοκότητες, ε, διατομιακές, ε, διεπιστημονικές ε, στην κοινωνία μας και θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση, να καταρτίζονται καλύτερα οι επαγγελματίες σε τέτοιου τομεί. Παραδείγματο χάρη, θα αναφέρω ένα παράδειγμα ιδιαίτερα πολύπλοκο με διασυνοριακό στοιχείο, το πώ καταπολεμούμε την νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, που είναι και προτεραιότητα τη νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλο, να αναφέρω ότι θέλουμε να τονίσουμε ότι αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να λάβει και υπόψη τις στενές σχέσεις που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με κάποιες τρίτες χώρες. Προσωπικά έχω εμπλακεί στο να παρακολουθώ το πώς αναπτύσσεται το δικαστικό σύστημα στη Μολδαβία, στη Γεωργία, στην Ουκρανία. Μέσω τέτοιων προγραμμάτων διασφαλίζουμε ότι και οι χώρες αυτές που είναι συνδεδεμένες με την Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη μπορούν τελικά να αγγιθούν την ορθή λειτουργία των δικαστικού του συστήματος και την ανεξαρτησία των δικαστών. Έτσι λοιπόν, διαθετήσω κάποιες από τις κριτικές που ακούστηκαν, αλλά νομίζω ότι κάποια άλλα στοιχεία θα συνεχίζουμε να τα υπερασπιζόμαστε. Σας ευχαριστώ. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ε, πιστεύω, θέλω να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές να επενθυμίσουμε την Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι η 5η Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Ολοκληρώνουμε τη σημερινή συνεδρίαση και θα ξεκινήσουμε αύριο στις 9 με τους συντονιστές και στις 10 έχουμε τις ψηφοφορίες. Ευχαριστώ πολύ όλες τις ομάδες προετοιμασίας και εργασίας και τους διερμηνείς.